το αίτημα αυτό ε, απεστάλησε στην Αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σας υποθυμερώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ελέγξαμε στην συνεδρίαση 21 Ιανουαρίου του 2013 της ε, ε, αρμοδιότητες και προτείναμε την κυρία Φραντσέσκα Μπαρατσιού από 17 Δεκεμβρίου 2012, τον κύριο Πρέσλαφ Μπορισόφ από 1η Ιανουαρίου 2013 και τον κύριο Ντομήτρου Σαμφιρέσκου από 9 Ιανουαρίου του 2013. Και σας προτείνω λοιπόν να επικυρώσουμε τις έντολες ε, αυτές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Μάλιστα, ε, έτσι επικυρώνονται οι εντολές αυτός. Ε, από τους μη εγγεγραμμένους ε, έλαβα έτοιμο ε,